σε σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων να μην υποβληθούν αντιρρήσεις για τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό που ανακοινώθηκε χθε στην έναξη της χθεσινής συνεδρίασης δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και ενστάσεις κατά το 24ωρο που πέρασε και σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 θεωρείται ότι εγκρίθηκε η σύσταση. Θα δημοσιευθεί με τα κείμενα που θα εγκριθούν για αύριο,